Ξεκινούμε με, την, ε, με τις αιτιολογήσεις ψήφου στην έκθεση Βαϊτσέκερ και το λόγο έχει για ένα λεπτό η κυρία Βον Στόχ. Κύριε Πρόεδρε, πρόκειται για τα εικονικά νομίσματα όπως τα bitcoin. Είναι πολύ θετικές οι επιπτώσεις που μπορούν να έχουν, δηλαδή εξοικονομήσεις ε, δισεκατομμυρίων. Πρόκειται για πραγματικά άλματα τεχνολογικά που επιτρέπουν ταχύτατες συναλλαγές μέσω του διαδικτύου. Αποκεντρωμένοι προσέγγιση όμως αυτή αποτρέπει οποιαδήποτε συγκεντρωτική εποπτεία και αυτό το πρόβλημα ενοχλεί τους γραφειοκράτες δεν ξέρουν τι να κάνουν απέναντι στην blockchain και αυτό το πνεύμα διακατέχει ολόκληρη την έκθεση όμως χρειαζόμαστε νέα τεχνολογία η οποία να μπορεί να λειτουργήσει και να αποδώσει χωρίς εποπτεία και επιτήρηση των γραφειοκρατών της Κομισιόν, της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας να μείνουν μακριά οι θεσμοί αυτοί από τα ε, ε, εικονικά νομίσματα. Ένα λεπτό, ο κύριος Μαμίκινς. Ε, Ευχαριστώ. Οι νομίσματα εμφανίστηκαν πριν από κάποια χρόνια όπως ε, τα bitcoins. Οι τεχνολογίες ε, σίγουρα επηρεάζουν σημαντικά τις ε, χρηματαγορές και άλλους τομείς, τις χρηματαγορές συγγνώμη, και άλλους τομείς και πιστεύω ότι πλέον θα πρέπει να αξιολογήσουμε το πώς αυτού του είδους τα νομίσματα ε, συνεισφέρουν ε, στην αγορά και πώς μπορούμε να ρυθμίσουμε τα σχετικά. Τα εικονικά νομίσματα μπορούν να περιορίσουν το κόστος των συναλλαγών, ιδίω των ε, διασυνοριακών μεταφορών πιστώσεων και θα μπορούσαν επίσης να χρησιμοποιηθούν και για την αρχιτεκτονική της ασφάλειας για να βελτιωθεί επίσης η ταχύτητα. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ και εγώ. Το λόγο έχει για ένα λεπτό ο κύριος Πόλτσακ. Děkuji, Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Θα συμφωνήσω με τους συναδέλφους μου και προσοχή, προσοχή να μην ενταχθούν στα ε, νομισματικά συστήματα, τα bitcoins και άλλα εικονικά νομίσματα χωρίς καμία απολύτως ε, εποπτεία. Δεν μπορεί κανείς ε, να ρυθμίσει κάθε ανθρώπινη δραστηριότητα, σε αυτό συμφωνώ. Όμω ενδέχεται κάτι τέτοιο να έχει σημαντικέ αρνητικέ επιπτώσει και αυτό είναι σημαντικό. Γι' αυτό θεωρώ ότι είναι καθήκον μα και καθήκον του νομοθέτου Ο μέγας φόβος είναι η νομιμοποίηση κερδών από οργανωμένη εγκληματική δράση και βεβαίως και η σημαντική αστάθεια που επιφέρουν τα, οικονομικά, τα εικονικά νομίσματα και με τις κερδοσκοπικές φούσκες οι οποίες μπορούν να οδηγήσουν σε κατάρρευση του συστήματος. Το λόγο έχει πάλι για ένα λεπτό ο κύριος Μαμίκινς. Κύριε Μαμίκινς, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Πριν από λίγα χρόνια ξεκίνησε η κρίση ε, με τους μετανάστες. Έχουμε δεχτεί στη χώρα μου τη Σουηδία πάνω από 300.000 αιτήσει για ένα εκατομμύριο πληθυσμό. Το υψηλότερο επίπεδο για ένα εκατομμύριο 30.000 πρόσφυγες, 11.000 συγγνώμη πρόσφυγες, το μεγαλύτερο δηλαδή ποσοστό σε σχέση με οποιαδήποτε άλλη ευρωπαϊκή χώρα. Ελήφθησαν οι αποφάσεις από το Συμβούλιο και με βάση αυτές θα πρέπει να δεχθεί 130.000 πρόσφυγες ε, σε άσυλο από την Ελλάδα και 430.000 ε, από την Ιταλία. Έχουμε ήδη λάβει όμως αρκετά. Ε, Ευχαριστώ. Το Δεκέμβριο του 2012 οι Σουηδοί ε, αμφισβήτησαν αυτό τον υποχρεωτικό χαρακτήρα των ποσοστώσεων όπως είχε συμφωνηθεί στο Συμβούλιο. Τελικά πάνω από 160.000 πρόσφυγες έλαβε το 2015, υποδέχθηκε το 2015 η χώρα και αυτό δημιούργησε έντονες πιέσεις ε, στο ε, σουηδικό σύστημα παροχής ασύλου. Δηλαδή δεν μπορούσαμε να δεκπεραιώσουμε όλα αυτά τα αιτήματα ε, διεθνούς προστασίας και από την άλλη πλευρά όλα τα κράτη-μέλη θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να δρομολογήσουν και το μηχανισμό προστασίας στην περίπτωση που έχουν να αντιμετωπίσουν κατεπίγουσες καταστάσεις, καταστάσεις εκτακτής ανάγκης όπως στην προκειμένη περίπτωση που έχουμε πολύ μεγάλο αριθμό του Ντονάσλο και άρχισε δεν μπορούν να το αντιμετωπίσουν. Ευχαριστώ. Με μεγάλη πλειοψηφία το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ε, εκφράστηκε ε, με την ψήφο του υπέρ της Σουηδίας ε, για να υπάρξει διακοπή ενό έτου, αναστολή ενό έτου, ό,τι αφορά το πρόγραμμα εγκατάσταση από την Ελλάδα στην Σουηδία. Εγώ είμαι μέλο του ΕΛΚΑ και αγωνίστηκα να αναγνωριστεί το γεγονό ότι η Σουηδία έχει λάβει, έχει υποδεχθεί πολλού περισσότερου ε, σε σχέση με άλλε χώρε ω χώρα υποδοχή. Είμαστε σε μια κατεπίδουσα κατάσταση, σε μια κατάσταση εκτακτή ανάγκη. Θα πρέπει λοιπόν να γίνει ένα προσωρινό διάλειμμα, αν θέλετε, να υπάρξει μια προσωρινή αναστολή ε, και βραχυπρόθεσμα ε, μόνο, διότι μακροπρόθεσμα θα μπορέσουμε ε, να συνεχίσουμε και στη Σουηδία να δεχόμαστε πρόσφυγες ε, με εξωπρεπή τρόπο. Η Σουηδία είναι μια ελευθερή χώρα, υπάρχουν ε, άνθρωποι οι οποίοι σίγουρα χρειάζονται βοήθεια και τους παρέχεται στη Σουηδία, αλλά θα πρέπει και άλλες χώρες ε, να βάλουν το δικό τους λιθαρακί. 28, ευχαριστώ. Και πάλι για την επόμενη έκθεση που αφορά το, το ψήφισμα που αφορά τις διατλαντικές ροές δεδομένων, ο κύριος Μαμίκινς. Κύριε Μαμίκινς, για τρίτη φορά εξηγήστε μας την ψήφο ε, Ευχαριστώ. Οι διατλαντικέ σχέσει σχέσει δηλαδή μεταξύ τη Ευρωπαϊκή Ένωση και των ΗΠΑ και του Κάναδα είναι οι πιο δραστήριε σε όλο τον κόσμο και έχουν και σημαντικό όγκο, οικονομικό όγκο. Τα δεδομένα δε είναι 15 τεραμπάιτ το δευτερόλεπτο. Ξεπερνούν όλες τις υπόλοιπες ανταλλαγές δεδομένων σε όλο τον κόσμο. Το 2014 η εισαγωγή ψηφιακών δεδομένων από την Ευρώπη ξεπερνούσε το 54% του συνόλου. Άρα πρόκειται για κάτι, για μια πτυχή δηλαδή από τις πιο σημαντικές στις διατλαντικές σχέσεις. Γι' αυτό το λόγο εγώ υποστήριξα την έκθεση. Ευχαριστώ. Την επόμενη εκθέση της κυρίας Γκρίφιν έχουμε τέσσερις επεξηγήσεις ψήφου. Ξεκινούμε με την κυρία Κίρτον Ντάρλινγκ. Για ένα λεπτό. Thank you, President. Energy poverty... Ευχαριστώ. Ενεργειακή φτώχεια ε, πλήττει πάνω από 50 εκατομμύρια στην Ευρώπη. Ε, που δυσκολεύονται να ε, εξασφαλίσουν τα προστοζήν και αυτό είναι απαρέδεκτο. Ένα στα δέκα νοικοκυριά πλήττονται στη δική μου περιφέρεια. Κανεί δεν θα έπρεπε να κλείνει το καλοριφέρ το χειμώνα. κανεί δεν θα έπρεπε να επιλέξει αν θα φάει ή θα ζεσταθεί. Καλωσορίζω την έκθεση ε, της Τέρεζα Γκρίφιν, εργατική συναδέλφου. Πρέπει τώρα να αναβαθμίσουμε τις προσπάθειές μας ε, να αντιμετωπίσουμε αυτά τα ζητήματα και ίσως να ληφθούν και μέτρα για την αντιμετώπιση των πραγματικών αιτίων της ενεργειακή φτώχειας. Οι καταναλωτές θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν την καλύτερη δυνατή λύση και ε, όχι ε, να αναγκαστούν να πληρώνουν τιμές που δεν τους συμφέρουν. Ψηφίσαν επίση κατά τις αυθέμητες εμπορικές κατά των αναθέμητων εμπορικών ε, πρακτικών και υπέρ συγκεκριμένων δράσεων για του πιο ευάλωτου ε, καταναλωτέ. Αλλά θεωρώ ότι μόνο με την έκθεση τη Τερέζα Γκρίφιν μπορούμε να προχωρήσουμε με σωστό τρόπο. Το λόγο έχει για ένα λεπτό ο κ. Μαμίκιν. Ευχαριστώ πολύ ε, αγαπητέ Πρόεδρε. Για την ώρα η Ευρωπαϊκή Ένωση βρίσκεται μέσα στη μέση μιας μεταρρυθμιστικής φάσης για την ενέργεια σε μια προσπάθεια αποκέντρωσης των συστημάτων παραγωγής ενέργειας αλλά και ε, βασισμένων σε ανανεώσιμες ενέργειες. Ο στόχος μας πρέπει να είναι να προσφέρουμε σταθερά μακροπρόθεσμα την ενέργεια ώστε και να ενισχύσουμε μάλιστα και τον κόσμο ώστε να μπορεί να παράγει και ο ίδιος ενέργεια δηλαδή οι ε, καταναλωτές οι ίδιοι και ιδίω σε πιο απομακρυσμένε περιοχέ. Βεβαίω και από την άλλη μεριά να έχουν δυνατότητα να επιλέγουν του προμηθευτέ του. Πιο μακροπρόθεσμα νομίζω ότι θα μπορέσουμε να απαναγούμε από τα μονοπόλια της ενέργειας. Σε ορισμένες χώρες αυτό παραμένει ένα πρόβλημα. η κυρία για ένα λεπτό. <clears throat> Ευχαριστώ. Το ενεργειακό σύστημα με την κεντρική θέρμανση είναι παρελθόν και θέλουμε πλέον να προωθήσουμε ένα σύστημα αυτό. Ο που θα στηρίζεται κυρίω και στις πηγέ πηγές ενέργειας. Ανακοίνωση τη Κομισιόν για τη νέα συμφωνία κατανάλωση ενέργεια. Ε, εδράζεται σε τρει πυλώνε. την καλύτερη ενημέρωση των καταναλωτών για να καταναλώνουν ώστε να ήταν λιγότερη ενέργεια και να δαπανούν βέβαια και λιγότερα χρήματα και βέβαια και άλλοι δύο πυλώνες, ε, περισσότερες επιλογές για τους καταναλωτές, ε, για παράδειγμα σε θέρμανσης και επίπεδο προστασίας των καταναλωτών, να είναι το, το, το υψηλότερο δυνατό. Αυτός είναι ο τρίτος πυλώνας. Επίσης, θα πρέπει να υπογραμμίσουμε τον ορισμό της ενεργειακής φτώχειας επίπεδο ένωσης, γιατί είναι τέλος διαφορετικές οι ανάγκες ενέργεια από τη μια χώρα στην άλλη και το ελάχιστο ε, εισόδημα κατά κεφαλή ε, επίσης είναι πολύ διαφορετικό από τη μια χώρα στην άλλη και τα κράτη επίσης αντιλαμβάνονται τελείως διαφορετικά την έννοια εύλογο κόστος. Όμως πρέπει να καταπολεμηθεί η ενεργειακή φτώχεια σε επίπεδο Ευρωπαϊκή Ένωση, για να μπορέσουμε να εφαρμόσουμε. Λόγο έχει για ένα λεπτό και πάλι ο κύριος Πόλτσακ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Εγώ υποστηρίζω το μέγα αυτό έργο της Ενεργειακής Ένωσης και τη δημιουργία μιας ενιαίας ενεργειακής αγοράς. Βεβαίως τα υποστηρίζω αυτά. Πρέπει όμως να είμαστε προσεκτικοί στον χώρο αυτό και να υπολογίσουμε προσεκτικά ποια μέτρα είναι εκείνα τα οποία πρέπει να κριθούν και να εφαρμοστούν στο ευρωπαϊκό επίπεδο και πια στο εθνικό. Αυτό είναι σημαντικό καθηκόν ιδίω για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η έκθεση λοιπόν που συζητήσαμε μου φαίνεται καλή και μου φαίνεται ιδιαίτερα καλό το ότι προσπαθεί να στηρίξει την ανταγωνιστικότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ε, επίσης βρίσκω σωστό το ότι ζητεί διαφάνεια στον τομέα της ενέργειας και κάνει την προσπάθεια να ιδρύσει μια πραγματικά ε, σωστά λειτουργούσα παραγωγή ενέργειας που θα επιτρέψει εν τέλος να προστατεύσουμε και τον κόσμο από τη φτώχεια. Τώρα στις δύο διευκρινήσεις ψήφου στην έκθεση της κυρίας Αρένα για τη φτώχεια μια προοπτική με γνώμονα το φύλλο. Ε, πρώτος έχει το λόγο ο κύριος Σκρίπεκ για ένα λεπτό. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Εδώ μιλούμε για τη φτώχεια των γυναικών, την ερική φτώχεια των γυναικών, δηλαδή τη διαφορά μεταξύ ανδρών και γυναικών. Και εδώ ε, ορίζονται διαφορετικές ανάγκες κάποιων ομάδων, ακόμη και μάλλον για τη φτώχεια κατά τον εξωτερικό Και πρέπει να ληφθεί υπόψη κατάσταση στη φτώχεια, στις ε, διαφορές αμοιβή μεταξύ ανδρών και γυναικών, διαφορές συντάξεων. Οι γυναίκες είναι φροντίστριες, φροντίζουν για ηλικιωμένους, παιδιά. Είναι επάλωτες ε, κάποιες κατηγορίες από αυτές, ε, ανήπαντρες, ε, αυτές που κινδυνεύουν να, ε, να χάσουν δουλειά τους, οι νεάνες κτλ. Θα πρέπει να καταπολεμήσουμε τη φτώχεια των γυναικών. αλλά όχι και να είναι διαφορετική αντιμετώπιση των γυναικών ε, ανάλογα το αν είναι λεσβίες ή δεν ξέρω αν ανήκει σε οποιαδήποτε άλλη κατηγορία ΛΟΑΔ. Εδώ μιλάμε για τις ε, γυναίκες ε, συγκεκριμένα. Αλλά θέλουμε να καταπολεμήσουμε τα στερεότυπα. Δεν μπορώ να στηρίξω όμως να φτάσουμε σε αυτό το σημείο. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. 64 εκατομμύρια γυναίκες και 57 εκατομμύρια ανδρών ζουν σε συνθήκες φτώχειας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο αριθμός των γυναικών λοιπόν είναι σημαντικά μεγαλύτερος. Επομένως το γυναικείο φύλλο υφίσταται περισσότερο τις δυσμενείς επιπτώσεις της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού. Για το λόγο αυτό πρέπει να τονίσουμε και το αποκρουστικό γεγονός ότι οι γυναίκες το βρίσκουν πιο δύσκολο να δραστηριοποιούνται επαγγελματικά για διαφόρους λόγους. Θα προτείνω λοιπόν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να εγγύψει το δυνατόν συντομότερο σε μια ε, συνολική στρατηγική που θα επιτρέψει να ικανοποιηθούν οι ανάγκες μητέρων, πατέρων. Ε, έχουν ειδικέ ανάγκες τα πρόσωπα αυτά. Ευχαριστώ. Έχουμε στην επόμενη έκθεση που είναι η έκθεση Ντάλτον δύο διευκρινήσεις ψήφου. Κύριε Μαμίκινς, μην κάθεστε, σηκωθείτε πάλι. Έχετε ένα λεπτό για διευκρινήση ψήφου. Ευχαριστώ πολύ. Αυτό που θα ήθελα να πω είναι ότι μετά τη μεταρρύθμιση νέας αγοράς, εδώ και 20 χρόνια, υπάρχει μια νέα αγορά. Χωρίς δασμολογικούς περιορισμούς, χωρίς δασμολογικούς φραγμούς, όμως τελικά υπάρχουν κάποιοι φραγμοί παρόλα αυτά. Καταλαβαίνουμε βέβαια ότι πρέπει να εξαλειφθεί στο βαθμό του δυνατού η γραφειοκρατία για την ψηφιακή αγορά μιλώ και θα πρέπει να βελτιθεί ποιότητα ε, των παρεχόμενων υπηρεσιών. Σε διάφορα κράτη-μέλη συχνά σε διαφορετικά συστήματα, οπότε προκύπτει η κατάσταση ότι παραδείγματος χάρη μια συστημένη επιστολή Το λόγο έχει για ένα λεπτό η κυρία Μακοβέη. Ευχαριστώ. Η δημιουργία κατέστη δυνατή επειδή υπήρχε ένας ενιαίος στόχος, δηλαδή η κατάργηση των φραγμών. Τώρα έχουμε ωστόσο φραγμούς μη δασμολογικού χαρακτήρα που οδηγούν ωστόσο σε επιβάρυνση, κοστολογική επιβάρυνση των επιχειρήσεων που επιθυμούν να βγουν στην ενιαία αγορά. Και αυτές πλήγονται περισσότερο. Και μιλώ για ρυθμίσεις ε, ΦΠΑ, για συμφωνίες μεταξύ ορισμένων χωρών μελών και κάποιων μεγάλων πολυεθνικών ομίλων. Αυτά όλα εγείρουν φραγμούς μη δασμολογικού χαρακτήρα που τελικώς αποβαίνουν σε βάρος των καταναλωτών. Η έλλειψη διαφάνειας, για παράδειγμα, για τις επιγραμμικές πωλήσει. Και αυτές αποτελούν φραγμούς μη δασμολογικού χαρακτήρα και μειώνουν την ανταγωνιστικότητα της ενιαίας αγοράς. Η τελειοποίηση της ενιαίας αγοράς με πλήρως ελεύθερες συναλλαγές θα αποφέρει σημαντικότατα κέρδη, άνω των 600 δισεκατομμυρίων. Η έκθεση όπου έχουν ζητηθεί επεξηγήσεις ψήφου είναι η έκθεση κόμη. Το λόγο έχει πάλι για ένα λεπτό η κυρία Μακοβέη. You have the floor again. Mrs. McAvey, you didn't ask. Okay. Δεν θέλει το λόγο, κυρία Μακοβέη, μάλιστα. Στιγμή που δεν θέλει το λόγο η κυρία Μακοβέη, ολοκληρώσαμε τις διευκρινήσεις ψήφου. Τα πρακτικά της ε, παρούσα συνεδρία, θα υποβληθούν στο σώμα προς έγκριση στην αρχή τη επόμενης συνεδρίασής του. Αν δεν υπάρχουν αντιρρήσεις θα διαβιβάσω τα ψηφίσματα που εγκρίθηκαν κατά τη σημερινή συνεδρίαση στα πρόσωπα και τους φορείς τα ονόματα των οποίων αναφέρονται στα ψηφίσματα. Η παρούσα σύνοδος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου διακόπτεται. Η συνεδρία